Άρχεται η συνεδρίαση. Οι αρμόδιε Ιταλικέ αρχέ με ενημέρωσαν για την εκλογή του κ. Τζοβάνι Μπαρμπαγκάλο. Η εκλογή του τίθεται σε ισχύ από τι 11 Μαρτίου του 2014 και ο κ. Μπαρμπαγκάλο αντικαθιστά την κυρία Μπαράτσο. Με βάση το άρθρο 7, παράγραφο 1 τη πράξη για τη διεξαγωγή απευθεία εκλογών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω επίση και με βάση το άρθρο 4 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση τη εκλογή του κ. Τζοβάνι Μπαρμπαγκάλο που τέθηκε σε ισχύ στι 11 Μαρτίου 2014. Χαιρετίζω, καλωσορίζω μάλλον τον νέο συνάδελφο και θέλω να επενθυμίσω ότι ο κ. Μπαρμπαγκάλο θα μπορεί να συμμετέχει ω πλήρε μέλο σε όλε τι συνεδριάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον βέβαια δεν έχει υπάρξει ένσταση εντωμεταξύ για την εκλογή του και εφόσον και ο ίδιο έχει δηλώσει σε γραπτή μορφή ότι δεν κατέχει άλλη θέση η οποία να βρίσκεται σε αντίθεση με τα καθήκοντά του του Ευρωβουλευτού. Ε, επί του διαδικαστικού, ο κ. Μποντί. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιρετικά περιστατικά και εξελίξεις που έχουμε στην γαλλική δημοκρατία, που πλήττουν ε, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Ε, πρόκειται για παραβίαση των ε, προσωπικών ελευθεριών. Πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην Υπουργή και νομική